Vážené ak dovolíte, začneme rokovanie Výboru pre práva žien a Ευχαριστώ και καλό απόγευμα σας. Καλώς ορίζω στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη την οποία έχετε λάβει. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι στην ημερήσια διάταξη. Όχι. Οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Επίσης ε, υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 5 και της 9ης ε, Μαρτίου στα εγγραφά σας. Ε, μέχρι το τέλος της συνεδρίας δεν έχει κανείς αντίρρηση. Υιοθετούνται και τα πρακτικά αυτά. Στην σημερινή μας συνεδρίαση έχουμε 19 γλώσσες στην διάθεσή μας, οπότε όλοι μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε τις γλώσσες σα μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Να σε ενημερώσω πως υπάρχουν εδώ υπάρχει και μια δημοσιογράφος ε, του BBC, η κυρία Βίλα, η οποία θα μαγνητοσκοπήσει την συνεδρίασή μας και η ψηφοφορία της κυρίας Λούλινγκ και η σχετική συζήτηση για την έκθεση Εστρέλα θα ε, συζητηθούν και βεβαίως ε, θα έχουμε και δύο προσκεκλημένους της κυρίας Φένσεν. Μιλάμε για καθηγητές ε, από το Όστοσον και το Σμέλεν της Σουηδίας, τους οποίους και καλωσορίζω στην ε, συνεδρίασή μας. Όπως ξέρετε θα είναι λίγο πιο σύντομη η σημερινή μας συνεδρίαση γιατί συνεδριάζουμε παράλληλα με την Επιτροπή Ήτρε θα κάνουμε μια κοινή ακρόαση με θέμα γυναίκες και επιστήμη. το δικό μας το κομμάτι θα ξεκινήσει 17 και 20 και θα χαιρόμουν να ολοκληρώσουμε άρα όσο τον πιο γρήγορα τις εργασίες μας. Και περνάμε τώρα σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Είναι οι ψηφοφορίες. Έχουμε δύο ψηφοφορίες σήμερα. Ως ε, συνήθως θα κάνω την ψηφοφορία στα γαλλικά. Έχουμε την έκθεση πρωτοβουλία της Επιτροπής Γυναικών με τίτλο Η μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα». Η συγγήτρια είναι η κυρία Λούλινγκ. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν πρόκειται για έκθεση πρωτοβουλίας. Είναι, μία, είναι μία από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είχαμε στα πλαίσια της συναπόφασης για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα. Πρόκειται για πολύ πολύ σημαντικό θέμα στα πλαίσια της συναπόφασης. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί μου και που κατέθεσαν τροπολογίες, καθώς και τις επιτροπές που κατέθεσαν γνωμοδοτήσεις. Σήμερα το πρωί συναντήθηκα με τον σκιώδη εισηγητή με τους σκιώδες συζητητές των υπόλοιπων ομάδων. Τους ευχαριστώ και για να σας διευκολύνω το έργο θα ήθελα να πω ότι έχουμε πολλές τροπολογίες για τον ορισμό των συντρόφων. Πολλοί συνάδελφοι έκαναν σχετικές προτάσεις. Εγώ θα ήθελα να παραμείνουμε στην, στον ορισμό που περιέχεται στην πρόταση της Επιτροπής, γιατί είναι ο πιο νομικά βάσιμος ορισμός. Αναφέρεται σε συζύγους ή συντρόφους ζωής που αναγνωρίζονται από το εθνικό δίκαιο. και οι οποίοι δεν είναι εταίροι της επιχείρησης ή μισθωτή της. Αυτός είναι ο ορισμός της προηγούμενης οδηγίας και δίνει το δικαίωμα στα κράτη-μέλη που δεν προβλέπουν συντρόφους ζωής να μην τους συμπεριλάβουν. Γιατί αναφέρεται σε εταίρου, σε συντρόφους με συγχωρείτε, που αναγνωρίζονται από την εθνική νομοθεσία. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσουμε όλοι επ' αυτού του ορισμού και να αφήσουμε κατά μέρος όλες τις υπόλοιπες τροπολογίες οι οποίες ουσιαστικά λένε το ίδιο πράγμα αλλά νομικά δεν είναι τόσο σίγουρες αν θέλετε. Και βεβαίως αυτός ο, ο ορισμός δεν χρειάζεται να μπει σε όλα τα σχετικά άρθρα όπως προβλέπουν πολλές τροπολογίες. Γιατί η δομή του κειμένου δείχνει ότι εφόσον υπάρχει ορισμός στην αρχή, αυτό ισχύει για όλο το κείμενο από εκεί και πέρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λούλινγκ. Με συγχωρείτε, δεν ήθελα να μειώσω ούτε τη σημασία της οδηγίας, ούτε την δική σας ε, σημασία ως εισηγήτριας. Η κυρία Γκρόνερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ, κυρία Λούλινγκ. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την τοποθέτηση της κυρίας Λούλινγκ ότι δεν πρέπει να έχουμε μια έκθεση η οποία δεν θα διαβάζεται. Συμφωνώ επίσης με το ότι οπωσδήποτε πρέπει να συμπεριλάβουμε τους συντρόφους και τις συντρόφους στην οδηγία, αυτό είναι το νέο σε αυτήν την οδηγία. Παρατηρώ όμως πως στις διάφορες γλώσσες υπάρχουν μεγάλες διαφορές οι Ισπανοί ε, συνάδελφοι κατέθεσαν μια τροπολογία η οποία έχει μεταφραστεί ως μόνο μέλη της οικογένειας, συγγενείς κτλ. Εδώ πέρα νομίζω μπορούμε να επανέλθουμε στον ορισμό της Κομισιόν και να πούμε θέλουμε οι σύντροφοι να συμπεριληφθούν ε, εκεί όπου αυτό προβλέπεται από την ομοθεσία των κρατών μελών. Επίσης ε, εδώ πέρα γίνεται λόγος ε, μόνο για συντρόφους συμβίωσης ε, άντρες ή γυναίκες. Αλλά υπάρχει και κάτι, μια άλλη διατύπωση άντρες και γυναίκες σύντροφοι συμβίωσης. Δεν ξέρω γιατί αυτή η επανάληψη αλλά η επανάληψη δημιουργεί και μία πολιτική διαφορά που δημιουργείται εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε τα πράγματα 20 φορές, οπότε νομίζω γενικά καλό είναι να ψηφίσουμε τους και τις ε, συντρόφους ε, στη χώρα η οποία το προβλέπει αυτό στην ομοθεσία της, αλλά οπωσδήποτε πρέπει μετά να δούμε ότι η μετάφραση είναι σωστή σε όλες τις γλώσσες γιατί δεν είναι ίδια η μετάφραση σε όλες τις γλώσσες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Αγκρένα. Κύριε Λούλινγκ, το καταλαβαίνω, γιατί ξέρετε, αλλιώ είναι σε κάθε γλώσσα. Στα γαλλικά και το αυθεντικό κείμενο είναι το γαλλικό κείμενο. Παίρνω την εκδοχή της Επιτροπής. Λέει, λέ partenaire de vie» Το λε στα γαλλικά είναι και τις και τους. Τώρα στα γερμανικά είναι partner κάθετος είναι. Γιατί έχετε αυτοαπασχολούμενους άνδρες και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες. Με άντρες αυτοαπασχολούμενους που έχουν σύντροφους άντρες ή γυναίκες και το ανάποδο. Αλλά το λέ στα γαλλικά είναι νομικά σαφές. Καλύπτει όλες τις πιθανότητες. Θα πρέπει να τονίσουμε ίσως στη μεταφραστική υπηρεσία ότι το κείμενο πρέπει να είναι σαφές και να καλύπτει άνδρες και γυναίκες. Και αυταποσχολούμενους και συντρόφους. Ευχαριστώ. Επτά, Το απολογία επτά της Επιτροπής Απασχόλησης, χωρίς αντικείμενο, δεν ψηφίζεται. Η επτά. άρχεται ψηφοφορία για το Σανζομπζέ. Περιμένω να βγάλετε τις κάρτες σας. No. Είστε έτοιμοι. Πέρας ψηφοφορίας. Τώρα ούτε η ψηφοφορία. Έχει την κάρτα της η κυρία Γκρένερ. Η κυρία Μαδουρέρ δεν έχει, αλλά τέλο πάντων η πλειοψηφία είναι τεράστια. απολογείο 8. Επιτροπή απασχόληση. έχει η ψηφοφορία. Για την 8. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ah oui, c'est rejeté. C'est 24. 25, 24. 25, 24 λέει η πρόεδρος. 28. Άρχεται, άρχεται η ψηφοφορία. Λεβοτεκλό. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 9. απολογία, ε, το απολογία της Επιτροπής Απασχόλησης και 4 της Νομικής Επιτροπής. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 10 και 2 τη επιτροπή Απασχόλησης. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 14 υπέρ 12 κατά εγκρίνεται. Το απολογείο 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 29. Και οι 5 της νομικής, γιατί είναι ίδιες. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11 της νομικής της Επιτροπής Απασχόλησης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. εννέα Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 31. Κατά τμήματα. Πρόεδρε, αφορά στον ορισμό, οπότε έχουν καταπέσει. Και αυτή έχει καταπέσει, 32. On vote maintenant l'amendement 12, la deuxième partie. Τροπολογία 12, δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέρας ψηφοφορίας. Rejeté. Απορρίπτεται. Το Υπουργείο 6 της νομικής άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 33. Άρχεται η ψηφοφορία. Oh, oui, Madame Το μικρόφωνο γίνεται. Ναι, μισό λεπτό. Προσπάθησα να εξηγήσω το πρωί την κατάσταση στους Shadow. Συμφωνήσαμε ότι η οδηγία αυτή αφορά κυρίως θέματα κοινωνικής ασφάλισης και την προστασία της μητρότητας για τους ανεξάρτητους. Ό, τους αυτοπασχολούμενους δηλαδή. Ό,τι αφορά αγωνικές άδειες θα περάσουν στην έκθεση Εστρέλα. Η τροπολογία της κυρίας Λάγκε είναι πολύ, η οποία μόλις ψηφίστηκε που είναι πολύ έξυπνη και που λέει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι μπορεί να έχουν άδεια όπως αυτή που περιλαμβάνει η οδηγία 92 είναι έξυπνο, παραπέρα δεν μπορεί να πάει. Η οδηγία 92 είναι αυτή όταν τροποποιηθεί θα αποφασίσει αν θα είναι γονική άδεια, άδεια πατρότητας, τι θα είναι. Εμείς παραπέρα ε, ψηφίσαμε μόνο το ότι έχουν ισότιμα δικαιώματα με τους ε, εργαζόμενους. Δεν την ήθελε εδώ γιατί δεν είναι εδώ η θέση της. Προσπάθησα να το εξηγήσω το πρωί στην κυρία Γκρένερ επί Μακρόν ότι δεν μπαίνουμε σε τέτοια ζητήματα εδώ. Γιατί προτείνω πρότεινα την υιοθέτηση της ε, τροπολογίας 35, εγώ απέσυρα την, ε, τις δικές μου για τις άδειες ε, μητρότητας και καλύπτουν όλες τις άλλες τροπολογίες. Ζητάμε να έχουν οι αυτοαπασχολούμενοι μετά από αίτημα και με την ευελιξία την ίδια άδεια. Και λέμε ότι απλά η άδειά τους δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό που αναφέρει η οδηγία. Αυτό που θα αναφέρει η οδηγία. Καλύψαμε τα πάντα. Γι' αυτό θα ζητήσω από την κυρία Γκρένερ να αποσύρει την τροπολογία της. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με την γονική άδεια και την άδεια μητρό, μητρότητας ή πατρότητας θα αντιμετωπιστούν σε άλλη οδηγία. Εγώ απλά με την τροπολογία 35 παραπέμπουμε στην, στο κείμενο αυτό παραπέμπουμε στην οδηγία. Η κυρία Γκρένερ. Κοιτάξτε για να μακρηγορούμε τώρα. Το σκεφτικό εδώ ήταν να συμπεριλάβουμε να δώσουμε τα ίδια δικαιώματα στους συντρόφους με τους συζύγους όταν το, το ζητήσουν. για να μπορεί να συμπεριληφθεί και να εγγυηθεί και η άδεια μητρότητας και η γονική άδεια και να μην αποκλείονται. Ευχαριστώ. Όχι, όχι, ο τίτλος είναι διαφορετικός εκεί στο 33. Λέτε μητρική άδεια και γονική άδεια. Άδεια μητρότητας και γονική άδεια. Επειδή αυτή η οδηγία αφορά μόνο την προστασία της ε, μητέρας, και εκεί πέρα συμπεριλαμβάνονται τα, τα πάντα τα υπόλοιπα στην έκθεση Εστρέλα. Ήθελα εδώ να μην μιλήσουμε γι' αυτό και να δεχτούμε την τροπολογία 35 όπου λέμε ακριβώς πως ε, τα δικαιώματα αυτά είναι τα ίδια με τις οδηγίες 29 και μετά έχουμε καλύψει τα πάντα. Αλλά περιμένουμε, δεν λέμε τίποτα εδώ πέρα για γονείς, ε, ε, για άδεια γονική πατρότητας και τα λοιπά. Και παραπέμπουμε στην άλλη οδηγία και ε, καλύπτεται και έχουμε και την ευελιξία. Με συγχωρείτε, αλλά ας μην ξανανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, ας ψηφίσουμε. Αν δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε, θεωρούμε ότι έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Γιατί ήταν ανοιχτή ψηφοφορία εδώ και ώρα. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 10 και 36 έχουν αποσυρθεί. 38. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτατα. 37 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζεται. Τέλος. Απορρίπτατα. Δεύτερο τμήμα. Ψηφίζεται παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτατα. 35. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η κυρία Λούλινγκ εκτός μικροφώνου λέει δεν δουλεύει η συσκευή μου. Βάλτε τη στη διπλανή. Τώρα δεν πρόκειται να λειτουργήσει γιατί έληξε ψηφοφορία. Είπαμε εγκρίνεται αυτή η τροπολογία. Η 34 καταπίπτει. Η 39 χωρίς αντικείμενο, η 13 χωρίς ψηφοφορία, 40 ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14 απασχόλησης. Πρώτο τμήμα. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην 14 της απασχόλησης, δεύτερο τμήμα. Ψηφίζεται τώρα. πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 41 καταπίπτει. 11. Ψηφίζεται. πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 42 καταπίπτει, 43 χωρίς αντικείμενο, 15 απασχόλησης χωρίς ψηφοφορία, 44 ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Για την 12 ψηφίζετε τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε τις 45. 7 της νομικής επιτροπής. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Κύριε Παναγιωτοπούλου. 13. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 8. 8 της νομικής. Ψηφίσατε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 14. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 9 της νομικής ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 15. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δέκα της νομικής ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 17 και 16 που είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 18. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 19. Ψηφίζετε. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 17 καταπίπτει 20. Ψηφίζατε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 1. Ψηφίζατε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 χωρίς αντικείμενο, 2. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 χωρίς αντικείμενο, 23. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Η 1 της έμπλη είναι χωρίς αντικείμενο. Ψηφίζουμε την 1 της νομικής επιτροπής. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 2 της νομικής επιτροπής. Ψηφίζεται παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Αν και οι σοσιαλιστές ψήφισαν υπέρ. Όχι. Όχι, με συγχωρείτε, εγκρίνεται, γιατί υπήρχε και μία ψήφος επιπλέον από τους σοσιαλιστές. Ψηφίζουμε τώρα την τρία. Ψηφίζετε παρακαλώ. πέρασε ψηφοφορίας. Κυρία Λούλινγκ. Εκτός μικροφώνου, κυρία Λούλινγκ. πέρασε ψηφοφορίας εγκρίνεται. Οι δύο έχει ψηφιστεί. 24 τώρα ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρία της νομικής. Καταπίπτει. Όχι. Ψηφίζουμε την τρία της νομικής επιτροπής. Ψηφίζεται τώρα. Πέρας ψηφοφορίας. Μικρόφωνο. Είχαμε την εντύπωση ότι ήταν η τρία της απασχόλησης. Αλλά εσείς εννοούσατε τρία της νομικής επιτροπής. Τότε είμαι κατά. να επαναληφθεί η ψηφοφορία γιατί νομίζαμε ότι ήταν η τρία της απασχόλησης, όχι της νομικής. Μπορείτε να επαναλάβετε την ψηφοφορία. Ωραία, επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Ψηφίζετε τώρα τρία της νομικής επιτροπής. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τρία της απασχόλησης. Έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέσσερα. Σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα, ψηφίζεται. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, ψηφίζεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Όχι, 25 καταπίπτει. Τροπολογία 4. Το πρώτο τμήμα είναι χωρίς αντικείμενο, δεν το ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα, τώρα. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα, χωρίς αντικείμενο. Το ίδιο ισχύει και για τις 5 και 6 της απασχόλησης. Περνάμε στην τροπολογία 26. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Τροπολογία 5. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 6. Ψηφίζετε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 27 είναι χωρίς αντικείμενο. Περνάμε στη τελική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίζεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Χωρίς καμία ψήφο κατά. Συγχαρητήρια κυρία Λούλινγκ. Κυρία Γκρένερ. Θέλω να, γραφτούν, να γραφτεί στα πρακτικά ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι μεταφράσεις για να συμπεριλαμβάνονται ε, άντρες και γυναίκες σύντροφοι και τότε συμφωνούμε. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστώ ξανά και συγχαίρω την εισηγήτρια κυρία Λούλεγκ. Δεύτερη ψηφοφορία έκθεση για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ισότητας γυναικών και ανδρών στο πλαίσιο των εργασιών των επιτροπών και των αντιπροσωπιών. Με εισηγείται την υποφαινόμενη. Να ζητήσω από την πρώτη αντιπρόεδρο, αλλά λέει η πρώτη αντιπρόεδρο ότι είναι αναγκαίο να αλλάξουμε την διεύθυνση των εργασιών. Να σας πω εξ αρχής ότι λίγο πριν το ξεκίνημα της ε, συνεδρίας είχα στείλει μια προφορική τροπολογία την οποία αποσύρω τώρα αλλά η κυρία δεν είχε αναγγείλει μια προφορική τροπολογία για την εννέα. Όταν φτάσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκρένερ. είστε έτοιμοι? Μες. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote Πέρας. Rejeté. Απολύπτεται. 7. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 8. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 9. Η κυρία Γκρένερ έχει εδώ την προφορική τροπολογία της. Ναι, για την τροπολογία που λέει ζητάει την δυνάμωση της λειτουργίας κτλ. λοιπά. Να μιλήσουμε και για τις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και η συμπλήρωσή μου και στα σώματα τα οποία ε, συστήνει το Κοινοβούλιο, όπως παραδείγματο χάρη αποστολές παρατηρητών εκλογών γιατί είναι και αυτή η άλλοι φορείς του Κοινοβουλίου, να υπάρχει και εκεί ισότητα. Euh, Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό. Δέκα. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία Εγκρίνεται. 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 13. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 14. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε. Λάθος. Ενιαία το ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή πρόταση. Η προσαρμογή καταπίπτει γιατί πέρασε η τροπολογία. Ομού τα τρία τελευταία. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Δεκτά. Ψηφίζουμε συνολικά το τελική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. δεκτή. Ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για τη συνεργασία σε όλους και όλες. teraz, dovolíte, prešli k e, bodu. A je to správa o... Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση σχετικά με το ταξίδι της αντιπροσωπείας στην Σουηδία. Θα πω εγώ λίγα πράγματα για το τι έκανε η αντιπροσωπεία μας και μετά ζητήσω από τους υπόλοιπους, τις υπόλοιπες συναδέλφους να κάνουν κάποιες παρατηρήσεις. Οι κυρίες Στρέλα, Σβένσον, Κοράτσο, Μπάουρ και Γκρένερ ήταν επίσης παρούσες στο ταξίδι αυτό. Το πρόγραμμα μας είχε συναντήσεις με μικαπαόμικρον, με προσώπους αρχών του κρατικού τομέα που ασχολούνται με την ισότητα. Επίσης συζητήσαμε με εκπροσώπους του Σουηδικού Κοινοβουλίου, με τον πρόεδρο, τον κύριο Βέστενμπεργκ και την κυρία Σκόνη, Υπουργό Ισότητας ανδρών και γυναικών, την κυρία Σένιο, τη Γενική Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, την κυρία Ζονγκατ, υφυπουργό του Υπουργείου Απασχόλησης, την κυρία Λίνο, η οποία είναι συνήγορος ε, για θέματα ισότητας, συνήγορος του πολίτη για θέματα ισότητας και τέλος ε, δώσαμε μια συνέντευξη τύπου και νομίζω πως όλες οι συνάδελφοι θα συμφωνήσουν μαζί μου στο ότι το σημαντικότερο θέμα των συζητήσεων ήταν το θέμα των εγγύων ε, εργαζομένων, εγγύων και ελεγχώνων. Ένα θέμα που ενδιαφέρει πολύ τους ε, Σουηδούς, και αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της Σουηδικής Προεδρίας. Διαφέρει λίγο η Σουηδική φιλοσοφία από τη δική μας ε, κατεύθυνση γιατί στην, από την ε, οδηγία μας μάλλον γιατί εκεί πέρα δεν είναι υποχρεωτική η άδεια μητρότητας και επαφίεται στον ή στην σύζυγο για το αν θέλουν αυτή την άδεια. Πρόκειται για μια άδεια 16 μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας η γυναίκα λαμβάνει 80% του μισθού της. Οι 16 αυτοί μήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το έκτο ε, έτος ηλικίας του παιδιού. Δύο μήνες είναι και για τους δύο γονείς ε, και τους υπόλοιπους μπορούν να τους μοιράσουν μεταξύ τους. Συναντηθήκαμε και με την συνήγορο για θέματα ισότητας, μια αρχή η οποία έχει αρκετά εκατομμύρια ευρώ προπολογισμό κάθε χρόνο, μια αρχή η οποία εφαρμόζει την Συμφωνία Περιμή μη διακριτικής μεταχείρισης. και οφείλω να πω πως η παρατήρηση και η επιτήρηση είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Είδαμε και το θέμα των ίσων αμοιβών. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την συνήγορο και οι υποθέσεις που έχουν καταδείξει, καταλήξει στα δικαστήρια. Είναι 5.500, 2.500 από αυτές έχουν κερδιθεί και βεβαίως ε, το κόστος αυτό είναι κάτι που θα επομιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Επίσης ε, το δίκαιο όσον αφορά την κατάληψη διοικητικών θέσεων είναι πολύ πιο προχωρημένο από τις άλλες χώρες Ευρώπης. Εκεί πέρα λοιπόν επενδύονται πολύ περισσότερα χρήματα στην ισότητα. Γύρω στα 400 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες ε, σε αυτή την θητεία της κυβέρνησης αντί για τα 40 εκατομμύρια που είχαν διατεθεί την προηγούμενη φορά. Επίσης ε, συζητήσαμε την ε, βία, την οικογενειακή βία, αλλά και την ε, πορνεία. Και υπάρχει και το σχέδιο δράσης κατά της πορνείας και της ε, εκμετάλλευσης των γυναικών της Σουηδικής κυβέρνησης και στο τέλος όπως σας είπα υπήρχε συνέντευξη τύπου νομίζω πως η κάλυψη στα μήμια ήταν πάρα πολύ καλή και εκπρόσωποι του Σουηδικού Κοινοβουλίου μας είπαν πως κατά διάρκεια της Προεδρίας θα έχουμε μία εκδήλωση, μία συνάντηση των δικτύων των Εθνικών Κοινοβουλίων και μας προσκάλεσαν και εμάς αυτή τη συνάντηση και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις συναδέλφους αυτής της Επιτροπής. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την κυρία Βεμπρίτση Σιλένσον για το ότι κύλησε καλά η επίσκεψή μας. Σας πολλές πληροφορίες για την προσοχή σου ειδική ε, προεδρία και να ευχαριστήσω και την κυρία Σφανέσταλ της Γραμματείας η οποία εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά για να είναι επιτυχημένο το ταξίδι αυτό της αντιπροσωπείας μας. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στις ε, συναδέλφους. Κυρία Μπάλα. E, Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, γεγονός είναι πως δεν υπάρχει στο Σουηδικό Κοινοβούλιο ανάλογη επιτροπή με την δική μας γιατί υπάρχει υπουργός και η συμμετοχή σε όλες τις επιτροπές. Επίσης, εάν οι φορείς εκεί της ισότητας κρίνουν υπέρ αυτού ο οποίο θεωρεί ότι υπέστη διάκριση, τότε δεν, ε, τότε δεν υπάρχουν δικαστικά έξοδα είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε νομίζω στο μέλλον. Είναι γνωστό πόσο πολλές περιπτώσεις διακριτικής ε, μεταχείρισης ξεχνιούνται γιατί βεβαίω ε, είναι και πολλά τα έξοδα. Και πραγματικά δεν είναι παντού ίδια η απόδοση και η νομοθεσία. Και το τρίτο το οποίο θα ήθελα να πω είναι η λύση της γονικής άδεια που είναι πολύ επίκαιρη για σχέση με την εκθεσία Στρέλα. Όσον αφορά το μέλλον, υπάρχουν κάποια προβλήματα διαδικαστικά, αλλά νομίζω πως καλό θα ήταν να εξυγχρονιστεί λίγο η προσέγγιση όπως και η οδηγία που πρέπει να ασχοληθεί λίγο και με την ασφάλεια. Πρέπει να δούμε λοιπόν το ζήτημα αυτό και να μπουν σε μία οδηγία και διαφορετικές αυτές άδειες. Αυτό είναι ένα από τα μαθήματα, ένα από τα διδάγματα αυτού του ταξιδιού. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνεισέφεραν για την οργάνωση αυτού του ταξιδιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Σβένσον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που συμμετείχαν ε, στην αποστολή. Θα ήθελα να πω στην Επιτροπή ότι μετά από αυτό το ταξίδι στην Σουηδία ασχοληθήκαμε με αρκετά ενδιαφέροντα θέματα. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια τώρα. Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας καλύφθηκε ευρέως από τα ΜΜΕ διαπιστώσαμε ότι σε σχέση με άλλες αποστολές η Επιτροπή μας έλαβε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη από ότι άλλες αντιπροσωπείες επιτροπών. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Σουηδοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την Επιτροπή μας στο Κοινοβούλιο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να παρακολουθούμε και εμείς τις εξελίξεις. Είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας, Και να προσθέσω κάτι όσον αφορά την πορνεία. Γνωρίζετε ποια είναι η Σουηδική νομοθεσία σχετικά. Συζητήθηκε αρκετά ειδικά οι διατάξεις που αφορούν την εμπορία ανθρώπων. Η Σουηδική κυβέρνηση οργάνωσε μία έρευνα για να διαπιστώσει ποιες είναι οι συνέπειες της υπάρχουσας νομοθεσίας για την πορνεία και την εμπορία ανθρώπων. Τέλος να πω ότι συζητήσαμε και το θέμα της γονικής άδειας. Πρόκειται για ένα σχέδιο οδηγίας που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Σουηδία. Συζητήσαμε λοιπόν εκτεταμένα το θέμα και θεωρείται ότι πρόκειται για μία οδηγία ελαχιστοποίησης. Αναφέρει τις ελάχιστες προδιαγραφές και από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη μπορούν να προχωρήσουν όσο περισσότερο θέλουν. Πρόκειται πάντως για μια οδηγία η οποία θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα όσα ισχύουν στη Σουηδία και προβλέπει υποχρεωτική άδεια για την μητέρα, κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει την αντιμετώπιση από τη Σουηδική νομοθεσία. Και Επαναλαμβάνω ότι χαίρομαι για, την, ε, για το ενδιαφέρον που δείξατε και ελπίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και για την Σουηδική Προεδρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τις συναδέλφους και να σας πω ότι η επίσκεψη ήταν και καρποφόρα και σημαντική, δημιουργώντας σοβαρότατο ενδιαφέρον από πλευράς των συνομιλητών μας <clears throat> και μικιό και μέλη του Κοινοβουλίου και μέλη της κυβερνήσεως αλλά και εκπροσώπους των μέσων. Προσωπικά θεωρώ ότι η Σουηδία είναι ένα κράτος μέλος όπου τα ζητήματα ισότητας παίζουν πολύ σπουδαίο ρόλο. Πρόκειται για μια χώρα που μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα. Ένα κράτος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως κράτος με βέλτιστες πρακτικές για την ισότητα ανδρών γυναικών. Γι' αυτό και η αντιπροσωπεία μας προκάλεσε τόσο ενδιαφέρον. Επίσης, τα θέματα που συζητώνται στην Επιτροπή μας αυτή τη στιγμή είναι θέματα που αποτελούν αντικείμενο των συζητήσεων στη Σουηδία. Ιδίως των συζητήσεων για την πρόταση οδηγίας για τη μητρότητα. Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω το εξή. Αυτό δεν αφορά τη Σουηδία, αφορά και άλλα κράτη. Πορτογαλία για παράδειγμα, την πατρίδα μου. Στην Πορτογαλία και αλλού βλέπουμε διαφορετικές καταστάσεις. Υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας και τη γονική άδεια. Υπάρχουν ωστόσο χώρες όπου η νομοθεσία καλύπτει όλους, όλες τις ε, πιθανότητες με έναν νόμο. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε βάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο που διακρίνει μεταξύ των διαφορετικών αυτών μορφών άδεια που καλύπτονται από διαφορετικές οδηγίες. Πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε ότι προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις άδειες σε μία οδηγία. Πρόκειται ωστόσο για μία σύσταση μόνο που μπορούμε να υποβάλουμε προς την Κομισιόν. Δεν έχουμε δικαίωμα πρωτοβουλίας, ε, νομοθετική πρωτοβουλίας στον τομέα αυτό. E Επιπλέον, πολλοί Συνάντησα πολλούς μεσογράφους στη Σουηδία και μετά από αυτά που είπε η κυρία Σφένσον θέλω και εγώ να υπογραμμίσω την αιτιολογική σκέψη 20 της οδηγίας που λέει ότι η οδηγία καθορίζει ελάχιστες ε, προδιαγραφές, επιτρέποντα όρους επιτρέποντας τα κράτη-μέλη να εισάγουν, να διατηρήσουν ευνοϊκότερες διατάξεις. Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν θίγει ούτε δικαιολογεί, δεν θίγει την υφιστάμενη κατάσταση, ούτε δικαιολογεί υποχώρηση της υφιστάμενης κατάστασης όπως ισχύει αυτή τη στιγμή στα κράτη-μέλη. Εμείς προτείνουμε λοιπόν ένα μίνιμουμ που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα. Πολύ διαφορετική. όχι μόνο σε ό,τι αφορά την διάρκεια των αδειών, αλλά και το κατά πόσον είναι ε, με αποδοχές ή χωρίς η άδεια αυτή. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι σε κανένα κράτος μέλος δεν υφίστανται οι πολίτες βλάβη λόγω της οδηγίας. Αν η εθνική νομοθεσία είναι ε, καλύτερη πιο Αυτό το λέει η αιτιολογική σκέψη 20. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το καταστήσουμε σαφές σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, ούτως ώστε να καταλάβουν ότι κανείς δεν θα βρεθεί σε μειονεκτικότερη θέση λόγω της εφαρμογής της οδηγίας αυτής. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν ότι πολλοί πολίτες θα κερδίσουν από την οδηγία αυτή. Στις χώρες όπου η νομοθεσία είναι λιγότερο ευνοϊκή αυτή τη στιγμή. Κύρια Κράτσα. Επιτρέψτε μου και μένα να σας συγχαρώ και σας προσωπικά που είχατε την ευθύνη και την ηγεσία αυτής της αποστολής, αλλά και τη γραμματεία που βοήθησε τους ώστε να γίνει ένα, ένα πρόγραμμα πλούσιο ενδιαφέρον και να πραγματοποιηθεί με μεγάλη ομαλότητα. Αυτά που θα ήθελα να επισημάνω συμπληρωματικά με αυτά που είπαν οι συναδέλφοι είναι ότι στη Σουηδία αντίθετα με άλλες χώρες το θέμα της ε, συμμετοχής στην πολιτική ζωή δεν αποτελεί μεγάλη πρόκληση διότι ε, όσο και να μην υπάρχει ισότητα απόλυτη παντού θεωρείται ένα θέμα λιμένο. Και αυτό α, ή με ποσοστώσεις ή με πολιτική οριμότητα και υπευθυνότητα όπως απήντησε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου είναι ένα θέμα το οποίο ε, έχει γίνει πρακτική καθημερινή. Ε, παρόλα αυτά όμως στη Σουηδία εξακολουθούν να τονίζουν οι υπεύθυνοι πολιτικά τις ε, ανισότητες που υφίστανται οι γυναίκες και ε, τόσο στην αγορά εργασίας όσο και ως θύματα της βίας. Και αυτό μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι όχι ότι η Σουηδία είναι μια χώρα ανισοτήτων ιδιαίτερα, αλλά είναι μια χώρα όπου το, όλη η, η, κουλτούρα, η κουλτούρα είναι τέτοια, η κοινωνική και η πολιτική, και η κοινωνική συνείδηση των ε, πολιτών τέτοια που καταγγέλλονται και επισημένονται οι ανισότητες, πράγματα που σε άλλες χώρες μπορεί να θεωρούνται ότι είναι φυσικό να συμβαίνουν. Ε, και αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα παράδειγμα ε, προς συζήτηση. Το άλλο που θέλω να πω, όπως αναφέρθηκε η κυρία Στρέλα, οι επεξηγήσεις που, που δώσαμε ότι η οδηγία, όπως και κάθε οδηγία, ε, αποτελεί ένα μήνυμο, είναι πολύ σημαντικό γιατί ίσως το, συναντήσουμε και για τις Σουηδέζες ε, συναδέλφους είναι σημαντικό στον προεκλογικό αγώνα να τονίσουν τι σημαίνει ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, και πώς πρέπει να, και πώς καλεί την αλληλεγγύη μας αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία για να εφαρμοστούν πράγματα σε κάποιες χώρες που δεν εφαρμόζονται καν ε, αλλά είναι και μια φορμή να δούμε και άλλα θέματα τέτοια πώς μπορούν να προκύψουν στον προεκλογικό αγώνα που οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν ότι μια οδηγία δεν είναι δυνατόν να τους οδηγήσει προς τα κάτω αλλά έχει σκοπό να οδηγήσει προς τα πάνω κάποιες χώρες που δεν έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο. Το άλλο που ήθελα να επισημάνω είναι την προετοιμασία που ήδη γίνεται και από την κυβέρνηση αλλά και από το Κοινοβούλιο ε, για την Σουηδική Προεδρία και μάλιστα ο Πρόεδρος μας είπε ότι ε, προετοιμάζει μια συνάντηση κορυφής τον Οκτώβριο με Προέδρους Κοινοβουλίων των, 27, των άλλων 26 χωρών, ελπίζω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπροσωπηθεί και άκουσε με ενδιαφέρον την πρόταση που του κάναμε στη συζήτηση, στην ατζέντα αυτή της συνάντησης κορυφής να ενταχθούν και η ανταλλαγή πρακτικών για την εφαρμογή της ισότητας. Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γκρένερ, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι αισθάνομαι ενισχυμένη για την πρόταση που έκανε η ομάδα μας για να πάμε στη Σουηδία για να δούμε την προετοιμασία της Σουηδικής Προεδρίας όσον αφορά την ισότητα και ήταν και η στιγμή επίκαιρη γιατί μπορούμε ακόμα να επηρεάσουμε, να κάνουμε ουσιαστικές συζητήσεις. Πάντα βεβαίως πάμε στη Σουηδία έχοντας κατά νου πως η Σουηδία είναι μία από τις πιο προχωρημένες χώρες στον τομέα αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιος είπε πως ε, ταξιδεύουμε στον παράδεισο στον παράδεισο της ισότητας και συναντάμε όμως μια πραγματικότητα ότι ακόμα και στην Σουηδία πολλά πράγματα είναι ακόμα στο στάδιο της επεξεργασίας και δεν είναι τέλεια. Γι' αυτό ήταν σημαντικό να δείξουμε στη Σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου ότι τα επιτεύγματα της Σουηδίας ε, που επιτεύχθηκαν βεβαίως ε, με το, το κοινωνικό κράτος που χρηματοδοτούν οι φορολογούμενοι σημαίνουν πράγματι ότι η Σουηδία έχει πετύχει να συμπεριλάβει τους άντρες στις δραστηριότητες ισότητας. Και οι άντρες ε, συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. 20% των Σουηδών πατεράδων παίρνουν ε, γονική άδεια για να βοηθήσουν και αυτοί στην ανατροφή των παιδιών. Και πραγματικά το βλέπουν και άσχημα και η κοινωνία το βλέπει και άσχημα εάν ένας πατέρας δεν ασχολείται καθόλου με τα παιδιά του. Οπότε έχει προχωρήσει λίγο περισσότερο η κοινωνία από άλλες χώρες. Γι' αυτό ήταν σημαντική αυτή η εμπειρία. Κάτι επί της ουσίας. Ελπίζω η Σουηδική Προεδρία να αναλάβει μια πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Σύνοδο των Γυναικών, να την αξιολογήσει καθώς θα έχουμε την πλατφόρμα του Πεκίνου που θα συμπληρώσει του χρόνου 15 χρόνια και χρειάζεται βεβαίως να γίνει απαραίτητη προετοιμασία Νομίζω έχουν ξεκινήσει ήδη οι Σουηδοί και τέλος, σημαντικό νομίζω ήταν, το ότι είχαμε επαφή με τα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, τον τύπο. Συνεισφέραμε να γνωστοποιηθούν και οι ευρωεκλογές στη Σουηδία. σε ευχαριστώ λοιπόν όλες ε, ήταν πραγματικά μια σημαντική και σωστή πρωτοβουλία. Ε, Ευχαριστώ την κυρία Γκρένερ. Να σας ευχαριστήσω, ευχαριστήσω όλες ε, τις συναδέλφους για τις παρατηρήσεις. Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση για την ε, βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία εγγύων λεχόνων και γαλουχουσών στο χώρο εργασίας. Από την ε, δημόσια ακρόαση και εδώ είχαμε αρκετές συζητήσεις και καταλήξαμε στις ε, τροπολογίες και νομίζω πως η συζήτηση θα είναι πολύ επικοδομητική και νομίζω πως ε, θα συζητήσουμε τις προτάσεις, αλλα... τις προτάσεις αλλαγής της πρότασης Εστρέλα, της τροπολογίες δηλαδή. Πρόκειται για μια έκθεση που αποτελεί αντικείμενο εργασία εδώ και πολλού μήνε και πλησιάζει επιτέλους το τέλος. Κυρία Στρέλα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροποποιήσεις και που συμβάλλουν σημαντικά στο κείμενο. Σίγουρα δε κάποιες από αυτές θα βελτιώσουν το κείμενο. Υποβλήθηκαν 107 προτάσεις τροποποιήσεις. Θα ήθελα να μιλήσω με, τους, με τις προτείνουσες και τους σκιώδεις εισηγητές για να πετύχουμε ε, κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Γιατί αλλιώ. Ε, όχι μόνο θα δυσκολευτούμε στην έγκριση, αλλά θα ενοποιημένες προτάσεις θα είναι πολύ πιο εύκολο να περάσουν στην Ολομέλεια. Είναι πολύ διαφορετικό να έχεις ε, μία πρόταση ή μία τροπολογία που να εγκρίθηκε με ομοφωνία στην Επιτροπή ή με μία πλειοψηφία οποιαδήποτε και να είναι. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω έκκληση στις συναδέλφους ούτω ώστε να με βοηθήσουν να βελτιώσω το κείμενο και να καταφέρουμε μία συνένεση που θα είναι θετική για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Εντάχει, θα ήθελα να σας πω ότι η διάρκεια της άδεια μητρότητα στον τομέα αυτό υπήρχαν πρωτοτροπολογίες που μιλούν για 14 εβδομάδες, κάτι που ήδη περιλαμβάνεται στην οδηγία του 92 και άλλες τροπολογίες που προτείνουν μια ε, διάρκεια 24 εβδομάδες. Μιλάμε δηλαδή για μια διαφορά 10 εβδομάδων μεταξύ των δύο προτάσεων τροποποίησης. Στην πρότασή μου προτείνω 20 εβδομάδες. Αλλά είμαι ανοιχτή. Και σε μια άλλη συμβιβαστική λύση που θα μπορούσε να γίνει δεκτή από τις περισσότερες σκιώδεις εισηγήτρες. Το πιο αμφιλογόμενο σημείο όπως ξέρετε, αφορά την ελάχιστη υποχρεωτική περίοδο της άδεια. Αυτό το είδαμε και στη Σουηδία. Η Επιτροπή προτείνει 6 εβδομάδες τουλάχιστον. Εγώ προτείνω 8. Οκτώ εβδομάδες μετά την γέννηση. Μετά το κεντό. Υπάρχουν όμως και προτάσεις που μιλούν για 2, για 4, για έξι εβδομάδες πριν και το αντίστοιχο μετά τον τοκετό. Υπάρχουν βλέπετε λοιπόν μεγάλες αποκλίνουσες απόψεις. Εγώ θα κάνω την μπορώ για να τα βρούμε. Για παράδειγμα, η κυρία Λούλινγκ προτείνει 8 εβδομάδες μετά τον τοκετό που μπορεί να επεκταθούν στις 12 κάποιες λένε υποχρεωτικά 16. Υπάρχουν του κόσμου προτάσεις δηλαδή. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια καλή ανάλυση της κατάστασης. γιατί ακόμη και η Σουηδία δεν κατάλαβα γιατί θέλουν να απορρίψουν μια διάρκεια που θα περιλαμβάνει έξι εβδομάδες πριν τον τοκετό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας λένε ότι έξι εβδομάδες είναι μήνυμο περίοδος για να μπορέσει η γυναίκα να πάει τα πάνω της μετά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Αυτό αποδεικνύεται δηλαδή επιστημονικά έξι εβδομάδες μετά τον τοκετό πρέπει να χρησιμοποιηθούν όπως και δίποτε από τη γυναίκα. Υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα φυσικής αποκατάστασης του σώματος και πρέπει η γυναίκα να μπορεί να χρησιμοποιήσει την άδεια αυτή. Μετά τις έξι εβδομάδες μπορεί η άδεια να μοιράζεται μεταξύ του συζύγου και του πατέρα μάλλον και της μητέρας. Και δύο μήνες να χρησιμοποιούνται από τον άντρα, δύο από τη γυναίκα. Συνολικά 8 εβδομάδες. Πιστεύω ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να το ξαναδουλέψουμε για να μπορέσουμε να, προσπε... να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Τώρα, για την συμπληρωματική περίοδο της άδεια. σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, γέννηση πολλών παιδιών, δι, διδήμων, τριδήμων κλπ ή γέννηση παιδιών με αναπηρίες ή γέννηση οκτώ μήνες μετά την προηγούμενη γέννηση. Περίπλοκες και σπάνιες περιπτώσεις που διαφέρουν από χώρα σε χώρα, εκεί πρέπει να έχουμε μια πιο ευέλικτη προσέγγιση. Πάντως, ε, η κατάσταση που αντιμετωπίζει η γυναίκα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική και άρα πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση πιο ευέλικτη. Τώρα γιατί την αμοιβή. Ε, εδώ νομίζω ότι υπάρχει, θα υπάρξει εύκολα συνένεση γιατί όλες οι προτάσεις έχουν ε, στόχο την καταβολή του 100% της αμοιβή της γυναίκας κατά τη διάρκεια της άδεια. Δεν πρέπει να επιβαρύνεται η γυναίκα επειδή γίνεται μητέρα. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναγνώριση των ίδιων δικαιωμάτων γονικής άδειας στις νέες μορφές οικογένειας, φερειπίν της ομοφιλόφιλες οικογένειες και εδώ μπορούμε να βρούμε μια συνέντευξη. Τώρα σε ό,τι αφορά ωστόσο την άδεια πατρότητας δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί. Να σας πω τα εξή, Ξέρετε ότι υπάρχουν προτάσεις που υπογραμμίζουν ιδιαίτερα την γονική άδεια. Υπάρχει μια οδηγία που ασχολείται ειδικά με την γονική άδεια. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε σε αυτή την οδηγία να συμπεριλάβουμε κάτι, ένα τομέα που ανήκει σε άλλη οδηγία. Γιατί αλλιώς δημιουργείται νομική σύγκρουση. Όπως ξέρετε, εδώ οι κοινωνικοί εταίροι έδωσαν την άποψή τους για τη γονική άδεια, συμφώνησαν και νομίζω ότι δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια που μας επιβάλλει η οδηγία. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, ε, χωρίς να έχω πλήρες, πλήρες δεν υπήρξε απόλυτη συμφωνία σε όλους τους ε, τομείς. Τώρα, για την άδεια πατρότητας, πρόκειται για μια σημαντική έννοια που πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ, γιατί χρειάζεται να κατανείμουμε τις ευθύνες μεταξύ των δύο γονέων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να υπάρξει ένας συμβιβασμός για την άδεια, για τη διάρκεια της άδεια πατρότητας. Σε ό,τι αφορά την κάλυψη όλων των εργαζομένων από την οδηγία αυτή. Σας ευχηστώ την προσοχή στο ότι η έκθεση που, που εγκρίναμε σήμερα της κυρίας Λούλινγκ αφορούσε τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε σύγχυση μεταξύ των δύο οδηγιών, νομικού χαρακτήρα κυρίως. Ως εκ τούτου, πρέπει στην οδηγία να συμπεριλάβουμε τις νοικοκυρές, αυτές που εργάζονται στο σπίτι και που δεν καλύπτονται από καμία οδηγία και προτείνω να καλύπτονται και οι εργαζόμενες και οι γυναίκες αυτές από την οδηγία. Να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογής της εργαζόμενες στο σπίτι. Για τις υπερορίες πιστεύω ότι μια συμφωνία θα υπάρξει εύκολα. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια συμβαστική λύση στο σημείο αυτό. Σε ό,τι αφορά την απαγόρευση απολύσεων, παρότι οι προτάσεις που έχουμε εδώ είναι τελείως διαφορετικές σε ό,τι αφορά την περίοδο προστασίας από πιθανή απόλυση, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Ίσως να μην συμφωνήσουν όλες οι ομάδες, αλλά πιστεύω ότι η πλειοψηφία των ομάδων θα συμφωνήσουν. Σε ό,τι αφορά τώρα τις άδειε θυλασμού. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις τροπολογίας, κυρίως μία για αγωνική, για περαιτέρω επέκταση της γονικής άδεια. υπάρχει μια για για περαιτερω επεκταση της γονικης άδειας. υπαρχει μια προταση που θέλει να εξασφαλίζει μείωση του χρόνου εργασίας για να μπορεί η μητέρα να πηγαίνει σε ιατρικές εξετάσεις. Θα πρέπει να δούμε μήπως αυτό προβλέπεται σε άλλες οδηγίες κυρίως, για παράδειγμα μάλλον, αυτή που ρυθμίζει την συμμετοχή των γυναικών και των ανθρώπων βέβαια στην αγορά εργασία. Μια άλλη πρόταση τροπολογίας αφορά την δημιουργία, την παρότρινση στη δημιουργία παιδικών σταθμών στους χώρους εργασίας, αποδεκτή νομίζω και άλλες τροπολογίες που προτείνουν να υπάρξουν κάποια φορολογικά κίνητρα για τους ε, εργαζόμενους. Καλή ιδέα. Η διατύπωση ωστόσο πάσχει κάπως. Συνολικά, όπως σας είπα, είχαμε 107 τροπολογίες που κατατέθηκαν από αύριο και μετά θα ξεκινήσω τις προσπάθειές μου να βρούμε συμβιβαστικές προτάσεις με τους συντάκτες και τις σκιώδεις εισηγήτριες για να βελτιώσουμε και την πρόταση της Επιτροπής και τις ιδέες που περιλαμβάνει η δική μου έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία εισηγήτρια. Τώρα θα ήθελα να ξεκινήσει η συζήτηση. Κύριε κυρία Φανλάνκη ζήτησε πρώτον λόγο. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και σένα Ιδίτ και αυτή την ωραία παρουσίαση των τροπολογιών. Θα ξεκινήσω με ζητώντα συγγνώμη για πολλές τροπολογίες μου και ο λόγος είναι απλός. Ξεκίνησα να γράφω με βάση κείμενα που δεν είχαν μεταφραστεί και σε διαβεβαιώ πως τα πορτογαλικά μου δεν είναι τόσο τέλεια ώστε να μπορώ να αντιληφθώ χωρίς λάθη αυτά τα οποία έγραφες εξού και αρκετές παρεξηγήσεις. Γι' αυτό συμφωνώ πράγματι πως θα είναι καλό εάν κάνουμε πράγματι κάτι για την ε, άδεια την εικονική, αλλά η δική σου η τροπολογία είναι πολύ καλύτερη από τη δική μου, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τις 100 ε, τροπολογίες. Αποσύρω την ε, δική μου. Πραγματικά λείπτει αυτή η διατύπωση όλες τις μορφές οικογένειες. Το ίδιο και για την 111 που αφορά τον θυλασμό. Πράγματι αυτό αναφέρεται στο 126 σε άλλη τροπολογία και είναι πολύ καλύτερα διατυπωμένο. Ε, στο τέλος απλά αναφέρεται στη δικιά μου πως θα πρέπει ο χρόνος αυτός να προσμετρηθεί ως χρόνος ε, εργασίας Είχαμε δύσκολη συζήτηση και ακόμα συνεχίζεται αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή για τον Υπολογισμό του Χρόνου Εργασίας και νομίζω πως πρέπει να πούμε ξεκάθαρα πως η περίοδος αυτή διακοπής ε, της εργασίας θα πρέπει να είναι μια περίοδος η οποία θα αμείβεται. Για τα υπόλοιπα πράγματι μιλάμε για επανένταξη και στήριξη στην εκπαίδευση των εργαζομένων για να μπορέσουν να επανέλθουν μετά από διακοπή της απασχόλησής τους ή να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί η διακριτική μεταχείριση. Λέμε λίγο πολύ ανάλογα πράγματα εκεί πέρα. Εντάξει, ίσως να είναι πιο θετικές διατυπώσεις από πλευράς κοινωνικού διαλόγου αλλά δεν νομίζω ότι διαφέρουν τόσο πολύ οι τροπολογίες μας, οπότε είμαι διατεθειμένη να βρούμε ένα συμβασμό. Μία συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να επισημάνω, το ότι η έγκυος γυναίκα πρέπει να έχει την ε, δυνατότητα να ζητήσει αλλαγή των ορών εργασίας της από τον εργοδότη αλλά τώρα υπάρχει το δικαίωμα να αρνηθεί κάτι τέτοιο ο εργοδότης αλλά θα πρέπει να πούμε πως θα πρέπει αυτή η άρνηση να είναι θεμελιωμένη και όχι να λέει απλά όχι. αλλαγή αυτή. Για τα υπόλοιπα καλή επιτυχία με τις συμβαστικές ε, λύσεις και ελπίζω να μην σε δυσκόλεψα. Πολύ ευχαριστώ. Mrs. Hannibal. Εκτός μικροφώνου. All right. <laughs> Sorry. Επιτέλους. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και σας ευχαριστώ και για την πολύ ολοκληρωμένη και επίκαιρη έκθεση. Είναι καλό που έχουμε μία νομοθετική πρόταση ως Κομισιόν για αυτό το θέμα που είναι τόσο σημαντικό για τις γυναίκες. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το όλο θέμα της ε, ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και κοινωνικής ζωής. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να υπάρξει πραγματική ισορροπία πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι άνδρες και να υπάρχει σαφής κατανομή των ευθυνών. Νομίζω ότι ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει αυτή η γυάλινη οροφή και δεν υπάρχει ίση πληρωμή είναι ότι δεν υπάρχει ίσως κατεμερισμός ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και όσο αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις δυνατότητες τους οι γυναίκες. Αυτό είναι λοιπόν που θα πρέπει να προωθήσουμε και δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε ακόμη και σε μικρή αύξηση της πατρικής άδειας. Το διαπιστώσαμε αυτό και στο Ηνωμένο Βασίλειο που πρότεινε την προηγούμενη εβδομάδα υποχρεωτική πατρική άδεια και υπήρξαν σημαντικές αντιδράσεις από πολύ κόσμο. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε. Είναι πολύ σημαντικό και είναι μια αρχή η οποία θα έπρεπε να είχε εγκαθιδρυθεί πριν από πολλά χρόνια και θα έχουμε τη δυνατότητα να την εγκαθιδρύσουμε με τη δική σας έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να γνωρίσω και εγώ το έργο της κυρίας Εστρέλα για τα όσα έκανε με αυτή την έκθεση. Να ευχαριστήσω και εγώ τους ε, συναδέλφους που κατέθεσαν τις 107 τροπολογίες. Λοιπόν θα ξεκινήσω από το τέλος. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα είναι το Μάιο, οπότε δεν υπάρχει ε, περίπτωση να εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Αυτό πιθανώς ενίσχυσε τον πειρασμό σε ορισμένους συναδέλφους να υπερβάλλουν γιατί θα παιχτεί και στην προεκλογική εκστρατεία αυτό το θέμα. Γι' αυτό είχαμε τις τόσες πολλές ε, τροπολογίες και κατατέθηκαν τόσες πολλές τροπολογίες που δεν έχουν και καμία σχέση τελικά με την οδηγία. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό αν είμαστε ειλικρινεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είμαι πεπισμένη πως αν συμφωνήσουμε πλήρως ε, πως πρέπει τουλάχιστον να σεβαστούμε τις πτυχές της υγείας που είναι πράγματι ε, αιτιολογημένες γιατί περί, αυ... περί αυτού πρόκειται θα ήθελα και εγώ να υποστηρίξω εδώ την εισηγήτρια. Απ' την άλλη θα ήθελα να ζητήσω κάτι από την γραμματεία. Προκειμένου η... Κοιτάξτε, επειδή μάλλον οι τροπολογίες ξεπερνούν τα πλαίσια αυτής της οδηγίας να τις επισημάνετε για να μην ψηφιστούν. Έτσι θα αποφευθούν πολλές παρεξηγήσεις πιστεύω. Είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό και το συζητήσαμε αυτό και την, στην τελευταία συνεδρίαση ότι δηλαδή το φθινόπωρο η Κομισιόν ε, όταν τελειώσει η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους σκοπεύει να καταθέσει μια πρόταση όσον αφορά την γονική άδεια και την άδεια πατρότητας. Οπότε είναι θέματα πέρα από το πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Ε, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι εκτός πεδίου ε, και θέλω να ζητήσω από την γραμματεία να προετοιμάσει μια ανάλογη λίστα. Ευχαριστώ κύριε Μπάουερ, κύριε Σφένσον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Εστρέλα για το έργο της. Πολύ ολοκληρωμένη η έκθεσή σας και πολύ σημαντικό το θέμα. Όσον αφορά τις τροπολογίες, έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα. Αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε είναι να καταλήξουμε σε κάποιες ε, χρήσιμες ε, συμβιβαστικές λύσεις. Είναι προφανές ότι εγώ και τα άλλα μέλη της ομάδας μου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να δείξουμε μια στάση αλληλέγγυα και να βελτιώσουμε τις συνθήκες για τις γυναίκες σε χώρες όπου δεν ισχύουν οι καλύτερες συνθήκες για την γονική και πατρική άδεια. Είμαστε φιλόδοξοι λοιπόν και θέλουμε να ισχύει ένα ελάχιστο επίπεδο για όλα τα κράτη-μέλη. Συζητάμε διάφορα θέματα ισότητας, ισότητα στο χώρο εργασίας και τα λοιπά. Μια βασική Προϋπόθεση όμως για την ισότητα είναι να δοθεί η δυνατότητα στις γυναίκες να καλύπτουν από μόνες τους τις ανάγκες τους και τις ανάγκες των παιδιών τους. Πέρα λοιπόν από θέματα ισότητας δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και τα δικαιώματα των παιδιών. περνάω στο θέμα των εβδομάδων της άδειας. Με βάση τις διάφορες προτάσεις που ακούσαμε από 18 με 24 εβδομάδες, θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό τελικά. Για την μητρική άδεια θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι θέμα ευθύνης της μητέρας από εκεί και πέρα. Γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε για ευθύνες έναντι του παιδιού που πρέπει να έχουν και οι δύο γονείς να μιλήσουμε για ευθύνη των γονέων οικειδεμόνων. Συμφωνώ με την εισηγήτρια και την σκιώδη εισηγήτρια που είπαν ότι έχουμε να κάνουμε με νομοθεσία του ελάχιστου. Δίνουμε τις ελάχιστες προϋποθέσεις και εγγύησεις και από εκεί και πέρα τα κράτη-μέλη μπορούν να προχωρήσουν περαιτέρω. Πώς λοιπόν θα βρούμε μία λύση στο πρόβλημα, αν διατηρήσουμε τη σύνταξη ως έχει, με υποχρεωτική μητρική άδεια για 8 εβδομάδες ας πούμε, αυτό θα έχει αντίκτυπο στην Σουηδική νομοθεσία για την γονική άδεια. Και θεωρώ ότι αυτές οι συνέπειες δεν θα γίνουν αποδεκτές από τους πολίτες της χώρας μου. Σήμερα προβλέπονται δύο εβδομάδες υποχρεωτικής άδειας για τις μητέρες. Αν περάσουμε σε 6-8 εβδομάδες, θα πρέπει η Σουηδία να αλλάξει την νομοθεσία της. Και δεν πρόκειται να υπάρξει ευνοϊκή υποδοχή αυτής της πρότασης. Τι θα κάνουμε λοιπόν με αυτό το πρόβλημα πολλοί αισθάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται με θέματα που δεν την αφορούν. Επαναλαμβάνω, θα υπάρξει πολύ αρνητική υποδοχή στην Σουηδία αν αλλάξετε την κατάσταση που ισχύει, ότι δηλαδή ο άνδρας και η γυναίκα από κοινού αποφασίζουν για το πώς θα μοιραστούν την άδεια. Εμείς στην νομοθεσία μας είχαμε ρυθμίσει το πρόβλημα. και αν υπήρχε πρόβλημα μετά την γένα, υπήρχε η δυνατότητα να λάβει η μητέρα ιατρική άδεια βασισμένη στην ασφάλιση ασθένειας που έχει. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την γονική άδεια, είναι επιπλέον. Άρα, στο θέμα της γονικής άδειας, το βασικό σημείο είναι τα δικαιώματα και η προστασία του παιδιού. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Και νομίζω ότι η φιλοδοξία όλων μας είναι να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα θέτει ελάχιστες προδιαγραφές προκειμένου όλοι να επωφεληθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, με συγχωρείτε η κυρία Φανλάνκε. Με συγχωρείτε. Ανησύχησα λίγο γιατί ενδιάμεσα ήρθε η κυρία Μπαν. θα ξαναξεκινήσω από την αρχή. Γιατί δεν... Το μήνυμα ήταν για σας. Ανησύχησα από τον ερχομό της κυρίας ε, Μπάουερ που ε, έδωσε εντολή στην γραμματεία. Συμφωνώ πράγματι πως οι εκθέσεις ε, που θα συνεχιστούν και στην επόμενη θητεία δεν πρέπει να είναι, δεν ξέρω, να κοτσάρει πάνω ό,τι θέλει ο καθένας μας. Αλλά το ότι μιλάμε και επιμένουμε τόσο πολύ για την υγεία και την ασφάλεια με ανισχύει βασίζεται και στην ισότητα. Οπότε μπορεί να είναι το εύρος λίγο πιο διευρυμένο από τις πτυχές μόνο της υγείας και της ασφάλειας της εγγύου γυναίκας. Δεν ανάγκη δηλαδή να ελέγχουμε και να διαλέγουμε τις τροπολογίες και να μείνουμε σε αυτές μόνο που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των χώρο και οι υπόλοιπε να φύγουν ανησυχώ γιατί σήμερα το πρωί κατά τη διεκαιάρκεια της ε, ψηφοφορίας στην Επιτροπή Εργασίας ο Φίλιππος Μάθιους, ο συντονιστής του ΕΛΚ, πήγε στην ίδια κατεύθυνση. Και φοβάμαι πως μετά από αυτά τα οποία έγιναν τις τελευταίες μέρες λάβαμε ένα, μια επιστολή από την Business Europe που έλεγε λίγο πολύ τα ίδια πράγματα. Δηλαδή να μην πούμε τίποτα σε αυτή την οδηγία για την καλύτερη κατανομή ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οπότε ζητώ από την ε, γραμματεία να λάβει υπόψη σοβαρά τις δύο νομικές βάσεις και να μην θεωρήσει ότι πρόκειται για μια δική που αφορά μόνο την υγιεινή και την ασφάλεια της χωροεργασίας. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Thank you very much, Mrs. Chair. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Στρέλα για το εξαιρετικό κείμενο εκθέσεώς της που περιλαμβάνει πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες. Όσοι ήθιστε προκατακτικά σχόλια θα κάνω, η Επιτροπή θα λάβει επίσημη θέση πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλεια να κάνω κάποια σχόλια ωστόσο για τις συζητήσεις για την ε, άδεια πατρότητα σε ένα από τα πιο καυτά θέματα. Ξέρουμε στην Επιτροπή ότι εσείς θέλετε να ενθαρρύνετε τους πατέρες να αποκτήσουν περισσότερες ευθύνε στην ανατροφή των παιδιών και συμφωνούμε μαζί σας. Ωστόσο δεν κάναμε τίποτα επί του θέματος γιατί οι κοινωνικοί εταίροι διαπραγματεύονται για τα θέματα γονικής άδειας και δεν ξέρουμε αν καλύπτεται και το θέμα της άδειας πατρότητας. Ε, πέτυχαν συμφωνία την περασμένη εβδομάδα, θα το εγκρίνουν ε, στο εσωτερικό του, των εταίρων, θα το στείλουν στην Επιτροπή και η Επιτροπή θα ετοιμάσει νομοθετική, νομοθετικό κείμενο βάσει αυτών των συμφωνιών, οπότε θα σας ενημερώσουμε. Ίσως είναι σημαντικό για τις συζητήσεις σας το εξή. Ένα από τα θέματα της συμφωνίας είναι ότι κοινωνικοί εταιροί πρότειναν να παραταθεί η γονική άδεια, γονική άδεια μιλάμε, κατά ένα μήνα. Από τρεις σε τέσσερις μήνες, εκ των οποίων ο ένας δεν θα είναι μεταφερόμενος. Ένας μήνας δηλαδή θα παραμείνει για τους πατεράδες. Αυτό αλλάζει την κατάσταση και πρέπει να το ξέρετε. Επίσης, ε, οι κοινωνικοί εταιροί δεν ασχολήθηκαν με το θέμα της άδειας πατρότητας. Θα λάβει υπόψη αυτό η Επιτροπή, θα λάβει υπόψη και το τι θα πει το Κοινοβούλιο και θα ε, λάβει απόφαση. Ελπίζω να ξεκαθάρισε τις διαφορές μεταξύ της γονικής άδεια για την οποία υπήρχε διαπραγμάτευση και συμφωνία των εταίρων και της άδεια πατρότητας που δεν εξετάστηκε. Αυτά θέλω να πω και να ευχαριστήσω εκ νέου την εισηγήτρια για την συνεργασία. Ελπίζω να υπάρξει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για την οδηγία. Ευχαριστώ. Merci Πέντε είναι. Τελειώνουμε κανονικά. Πολύ σύντομα. Τρία πράγματα να σας πω. Ένα. Το πολιτισμικό πρόβλημα. Η διαφορά νοοτροπίας. Και πρακτικών που ήδη υπάρχουν στα κράτη. Σε κάποια κράτη αλλά όχι σε άλλα. Με την οδηγία και τις τροπολογίες θέλουμε να βελτιώσουμε την κοινοτική νομοθεσία για όλα τα κράτη, χωρίς να επηρεάσουμε τα κράτη όπου έχουν ευνοϊκότερη νομοθεσία. Αυξάνοντας λοιπόν τα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών και χορηγώντας ευθύνες και στους δύο για να μοιράζονται την ευθύνη του γονέα. Για παράδειγμα, στη Σουηδία, καλός πατέρας δεν είναι αυτός που δεν χρησιμοποιεί την άδεια πατρότητας. Αντίθετα, στη Νότια Ευρώπη, κάποια κράτη, σε κάποια κράτη, ο πατέρας που παίρνει άδεια πατρότητας γελιοποιείται στη δουλειά του. Θέλουμε λοιπόν άδεια πατρότητας υποχρεωτική, ούτως ώστε αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την άδεια αυτή να μην τους δουλεύουν οι συνάδελφοί τους. Αυτά που είπε η κυρία Μπάουερ. Διευρύνεται η νομική βάση της οδηγίας, αλλά η εισαγωγή του άρθρου 140 της συνθήκης για την ε, προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί νέα βάση που μας επιτρέπει να εισάγουμε την έννοια της πατρότητας, προωθώντας έτσι την ισότητα φίλων. Άρα, τα θέματα υγείας του ατόμου δεν είναι δεν αποτελούν τη μόνη νομική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται πλέον η οδηγία. Αυτά που είπε η κυρία Σβένσον τώρα. Οι γιατροί τι λένε στη Σουηδία. Ίσως οι γιατροί δεν θεωρούν ότι για την ε, λεχόνα χρειάζεται μία μίνιμουμ περίοδος για να ανακτήσει τις δυνάμεις της η γυναίκα. Ο τοκετός δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ασθένεια. Είναι κάτι φυσικό. Πλην όμως απαιτεί να μπορέσει η γυναίκα να πάει τα πάνω της. Εγώ είχα αντίστοιχε συζητήσει με γυναικολόγους, με, με Όλοι μου είπαν ότι οι γυναίκε χρειάζεται, χρειάζεται μια, έναν επαρκή χρόνο για να αποκατασταθεί η υγεία της και μιλούν για έξι εβδομάδες. Δεν είναι προσωπική επιλογή του ατόμου, αλλά προστασία της υγείας της γυναίκας. Το αναφέρει άλλωστε αυτό το αναφέρουν αυτό και οι διεθνείς οργανισμοί και οι ειδικοί. Όλοι. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνεται λόγος για επέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα όταν μας αρέσει, όταν δεν μας αρέσει κάτι, μετά να φωνάζουμε ότι μπαίνει στα χωράφια τα εθνικά η Επιτροπή έλεος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για παράδεκτη επέμβαση στην ε, προσωπική ζωή του ατόμου. Βάσει των πληροφοριών που έχουμε, επεκτείνεται, διευρύνεται η άδεια μητρότητας ή υπατρότητας, όχι ωστόσο η αμοιβή. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα και αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία εύχομαι. Με την ολοκλήρωση εκεί της έκθεσής σας. Σας ευχαριστώ όλους ως κατές ανθρωπολογίες. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 16 Τετάρτου και στην ε, Ολομέλεια του Μαΐου. Στην τελευταία δηλαδή Ολομέλεια αυτής της ε, θητείας. Σας ευχαριστώ όλους και σας προσκαλώ στην συνέχεια της δημόσιας ακρόασης που βρίσκεται. Σας προσκαλώ λοιπόν στην ε, δημόσια ακρόαση στην PHS 1α02 και να σας ανακοινώσω πως η επόμενη συνεδρίαση είναι την 5η 16 Απριλίου από τις 9 μέχρι τις 11. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους διερμηνείς.